Ενημέρωσαν για την εκλογή του κυρίου Χάνου Τακούλα που αντικαθιστά τον κύριο Λιρέν από τις 27 Απριλίου του τρέχοντος έτους. Καλωσορίσατε, συνάδελφε και σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού και ενώ οι ε, αρμοδιότητες του δεν έχουν επαληθευθεί και δεν έχουν αποφασιστεί, ο κύριος Χάνου Τακούλα ε, ε, δρεύει με πλήρη δικαιώματα στο Κοινοβούλιο και στα όργανα του γιατί δήλωσε ότι δεν, δεν ασκεί καμιά άλλη ασύμβατη θέση, λειτουργία ασύμβατη με το λειτουργήμα του Ευρωπαϊκού